Possiamo iniziare i nostri lavori, questa aula molto grande, Λοιπόν, έχουμε σκορπίσει λίγο γιατί είναι μεγάλο ο χώρος. Λοιπόν, έχει διανεμηθεί το σχέδιο ημερήσιας διάταξης από τον Ιούλιο. Ένα πράγμα έχουμε να κάνουμε σήμερα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, το κομμάτι που μας αναλογεί. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές αν μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής θα μπορούσαμε να κάνουμε μία συνάντηση των συντονιστών. Σύντομα θα έλεγα, θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποια σημαντικά θέματα και να τελειώσουμε όλα όσα έχουμε να κάνουμε πριν από τις 1 και 4 που φεύγουν οι διευμηνείς. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρείται δεκτή η μερίσια διάταξη. Πριν περάσω στην ψηφοφορία, θυμίζω ότι είναι σαφές, πλέον πλησιάζει η επίσκεψή μας στην Ιταλία. Την προγραμματίζουμε εδώ και καιρό. Εδώ καλωσορίζω και την κυρία Κούρμαη, από τις 19 μέχρι 21 Οκτωβρίου θα γίνει η επίσκεψη στην Ιταλία. Παραμένουμε την άδεια, αλλά είναι προφανές ότι θα μας τη δώσουν. Προβλέπεται μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν πρόεδρος αυτής εδώ της Επιτροπής. Η συνάντηση αυτή θα γίνει το πρωί της 21ης Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας στις 19, όχι στη Ρώμη, αλλά στη Φλωρεντία γιατί θέλουμε να επισκεφθούμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Ήδη συζήτησα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου, θα γίνει μια συνάντηση με τους φοιτητές και ίσως και με τους καθηγητές, δεν ξέρω αν θα γίνει από κοινού ή ξεχωριστά. Έχουμε μια πρόσκληση πάντως από πλευράς του Ινστιτούτου να διπνήσουμε στο Ινστιτούτο αυτό που βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος με τρομακτική θέα πάνω από την πόλη της Φλωρεντίας <coughs> και αυτό θα μας επιτρέψει να παράσουμε καλά. Το πρωί της 20ης του μηνός θα φύγουμε για τη Ρώμη και θα έχουμε τις προβλεπόμενες συναντήσεις με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής και της Γερουσίας και στο τέλος, το απόγευμα της ίδιας μέρας, θα έχουμε θεσμικές συζητήσεις με υπουργούς και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Αν είναι δυνατόν το πρωί της επόμενης μέρας θα συναντήσουμε και τα μέλη του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου ή τουλάχιστον τον πρόεδρο του. Δεν έχουμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Θα δούμε αν μπορούμε να οργανώσουμε το ίδιο το πρωινό ή το προηγούμενο απόγευμα με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η αντιπροσωπεία εκτός από ΜΕ θα προσωπεύεται από τρία μέλη του ΕΛΚΑ, δύο των σοσιαλιστών και έναν από όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες. Δεν ξέρω αν έχουν ήδη οριστεί τα μέλη, για το ΕΛΚΑ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εδώ, Μέντες, α, εδώ είναι, μαζί μας είναι. Δεν μπορώ να σας δώσω ονόματα σήμερα ή θα κάνουμε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα και θα σας ενημερώσω. Την επόμενη εβδομάδα για τους σοσιαλιστές έχουμε ήδη τον Γκουερέρο, Γκουαλτιέρη. Για τον Γκουερέρο πρέπει να τον συγχαρούμε ότι είναι και με, ε, περιπτώσει, είναι μια χαρά και τον συγχαίρουμε για την του εδώ. Και υπάρχουν και άλλοι βουλευτές από δύο πολιτικές ομάδες, αλλά δεν έχουμε το όνομα άλλων δύο πολιτικών ομάδων. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω καμιά άλλη ανακοίνωση. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στις ψηφοφορίες για το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Πρώτα θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες που προτείνουμε στον προϋπολογισμό και μετά στη θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού. Και στο τέλος τη δική μας νομοδότηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο εισηγητής, ο συνάλφος Σαουντάργκας θέλει να εκφράσει την άποψή του, έχει την δυνατότητα να το κάνει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια αύξηση της χρηματοδότησης κάτω από τις τωρινές συγκυρίες. Είναι εντάξει με τη διερμηνία. Υπάρχει ένα συνεχής βόμβος. Ar, ar, ar girdite? Viskas gerai? O. pirmininkė, e, e, labai trumpai tik tai pasakyti, kadangi... Θα ήθελα λοιπόν εν συντομία να σας πω. Είναι εντάξει τώρα. Ναι, ναι, τώρα είναι εντάξει όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Επομένως, <clears throat> εν συντομία ήθελα να σας πω ότι κάτω από τις ε, τωρινές περιστάσεις δεν μπορούμε να προσδοκούμε μεγάλες αυξήσεις στα κονδύλια. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη το συμβολικό χαρακτήρα ορισμένων τομέων που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και χαίρομαι πολύ που υπήρξε και συνένεση μεταξύ όλων των συναδέλφων και μπόρεσα να συμπεριλάβω όλα τα σχόλια των συναδέλφων, εκτός από μια περίπτωση όπου θεωρώ ότι η διατύπωση του συναδέλφου ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υποστηρίξετε την θέση μου και ευχαριστώ. Μπαίνει. Πολύ ωραία. Θέλει κάποιος άλλος ε, να σχολιάσει. Όχι. Επομένως μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία τροπολογίες άμεσες για το γενικό προϋπολογισμό όλα τα τμήματα. Έχουμε εννέα τροπολογίες τέτοιες. Αναρωτιέμαι, ε, έχουν υποβληθεί από διάφορους βεβαίως ε, ε, από διάφορους συγγραφείς. Αναρωτιέμαι όμως εάν μπορούμε να ψηφίσουμε on μπλόκ τις τροπολογίες αυτές. Να ψηφίσουμε μία προς μία τις τροπολογίες. Εντάξει. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 6958 Κουρμάι και Γκερέρο υπέρ υπέρ εγκρίνεται νομίζω δεν υπάρχει κανείς κατά 1956 sempre proposto da e Ψηφίζουμε τώρα την 6956 και Γκερέρο υπέρ κατά Τέσσερις ψήφοι, κατά, όχι, πέντε. Εγκρίνεται πάντως. Τροπολογία 69-59, πάντα τον Κουρμάη και Γκερέρο. Υπέρ. Α, όχι. Έχει καταπέσει. Όχι, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε κανονικά 69-59 υπέρ. κατά εγκρίνεται με δύο ψήφους κατά. Επομένως δεν θα ψηφίσουμε την επόμενη τροπολογία, την 6950 δηλαδή. Ψηφίζουμε τώρα την 6951 του εισηγητού υπέρ κατά τρεις ψήφοι κατά, πάντως εγκρίνεται. Τροπολογία 6954, Χέφνερ, υπέρ. Κατά. Καμία ψήφος ε, κατά. Τροπολογία 6952 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6955. Χέφνερ. Υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6953 Γκερέρο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, όχι, μάλλον με δύο ψήφους ε, κατά. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες επί, τις τροπολογίες επί της γνωμοδότησης. Τροπολογία 1. Γέτερ Μάνκι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Γκερέρο. Υπέρ. Κατά. Τροπολογία 3. Γκερέρο. Υπέρ. Ε, κατά. Πέντε ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Επομένως, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην τελική ψηφοφορία ε, του, της τροποποιημένης γνωμοδότησης υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και Μία αποχή. Και μία αποχή. Πάρα πολύ ωραία. Άψογα. Στην ουσία δηλαδή τώρα σχεδόν τελειώσαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Μένει μόνο να πω ότι θα ξανασυναντηθούμε την ε, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στις 3 μέχρι τις 8.30, μέχρι τις 6.30 συγγνώμη και στις 5 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 στις Βρυξέλλες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας και παρακαλούνται οι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα.